Ελπίζω να έχετε όλοι τις ηλεκτρονικές σας κάρτες, γιατί όταν είναι μικρή διαφορά, δεν χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση κάθε φορά. Λοιπόν, αρχίζουμε. Σημείο 7. Συντονιστές είναι το 7 όχι, οκτώ. Βιομηχανικές εκπομπές. Η έκθεση Holger Kramer. Έχετε τον κατάλογο ψηφοφορία ε, στα χέρια σας. Και έχουμε και ένα συμβαστικό πακέτο. Πρώτο-πρώτο. Βλέπετε, καλύπτει πολλές ε, τροπολογίες. Και σας ερωτώ ποιος είναι υπέρ του συμβιβαστικού πακέτου. Ψήφι υπέρ, παρακαλώ. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ωραία, αυτό μας διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή για τις επόμενες ψηφοφορίες. Συνεχίζουμε. Η εννέα του εισηγητού ψηφιπέ Κατά. Enthaltungen angenommen. Ε, αποχές εγκρίνεται. Η 83. Ψήφι πέ. Dagegen. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ. Dagegen. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. παριθμόν 10 τώρα του εισηγητή. Α, έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Τμήμα πρώτο είπε. Κατά. Αποχές. κρίνεται. Το δεύτερο είπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλλά ας το ελέξουμε. Τσεκ το δεύτερο τμήμα. Τσεκ. Δουλεύουν τα μηχανήματα. Λοιπόν, αρχίζει ψηφοφορία, το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε τις ε, τροπολογίες βαριθμών 10. Abstimmung beendet. Πέρας. Α, ήταν σαφέ τελικά. 9 υπέρ, 31 κατά. Απορρίπτεται. Έχουμε δύο ταυτόσημες, 85 και 86 τώρα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαριθμών 87 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ. Για την 87. So, beendet. Peras. Peras. Α, εδώ όμως ήταν η μικρή διαφορά. 23 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται η 87. Τώρα έχουμε την 88 και την 89 που είναι ίδιες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 90 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφτεται. Η 11 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Identisch 92 94 είναι ίδιες. Όχι. Όχι, καλά. 92 και 93 ψήφι υπέρ. κατά απόχες απορρίπτεται τσεκ καλά Beendet. Πέρας. 28 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. Και 92 και 93 επευκαιρία. Λοιπόν, καταπίπτει τώρα 94 και πάμε στην 95. Ψήφι πέ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Check χωρίς την 95. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Beendet. Λοιπόν, απερίφθη όπως το είχα δει εγώ, 23 υπέρ, 27 κατά. 96 ψήφι υπέρ. Κάτα. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 98 και 99 είναι ίδιες ψήφι υπέρ. Όχι, πρώτα την 97 πρέπει να ψηφίσουμε, λέει. Ε, υπέρ. 97 Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 98 και 99 είναι ίδιες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ή 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 100 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα συνεχίζουμε σελίδα 5 παρακαλώ. Έχουμε τις τροπολογίες 117, 18 και 19 που είναι οι ίδιες και οι τρεις αυτές. Ψήφι υπέρ. Κατά. Όποχες. Εγκρίνονται. Οι 120 ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνονται 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121. 122. 123. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται, αλλά σας ελέγξουμε καλύτερα. Γιατί 121, 22 και 23 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Abstimmung beendet ναι, εδώ ήταν όντως μικρή διαφορά, ισοψηφία δηλαδή, απορρίπτεται 25-25. 124 äh, είναι παράδεκτη και πάμε στην 20. Το εισηγητή, ψήφιπε. Κατά Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 126 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, τώρα γυρίστε πολλές σελίδες μέχρι που... Α, μέχρι την 11. Κάτω, κάτω. 23 του εισηγητή. Ψήφιπε. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για την 23. Εγκρίθηκε με μικρή διαφορά 26-24. 165. Ψήφι πέρα. κατά αποχές απορρίπτεται. 24 ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 είπε, Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ορίστε. Τσεκ. Καλά. 27. Ας την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Ορίστε. Ε, είναι σαφές. 32 υπέρ, 22 κατά. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά αποχές Απορρίφτεται. 167 υπέρ κατά αποχές Απορρίφτεται. 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 τώρα ψήφι υπέρ 171. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 175-76 μαζί υπέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 174 έχει αποσυρθεί. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 178, 79, 80 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρα. Α, εντάξει. Απερίφθη σαφώ 22 υπέρ, 33 κατά. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές από 182-84 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τσεκ. <coughs> Καλά. 182-184 τις ελέγχουμε. πέρασε Εγκρίνεται 31 26. Ορίστε. Εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε. 185, 186, 187, 188 ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος παρακαλώ. Abstimmung beendet. 27 υπέρ, 29 κατά. Όπω σα είχα πει, απερίφθη. Αυτό είχα δει εγώ. Πάμε στην 191. Ψήφι υπέρ. Τη 191. Κατά. Αποχές. Απορρίψτε. 193 υπέρ. Ρώση. Α, ο ίδιος ο συντάκτης είναι κατά, ε, καλά. Ε, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Καταψηφίζετε την ίδια σας την τροπολογία. Ναι. Καλά. 192 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 194 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι απερίφθησης, αλλά στον έξω. 195. Πέρας. Mm, απερίφθη όντως. 195. 27 υπέρ, 29 κατά. 196 υπέρ. Κατά. Απόχες ε, εγκρίνεται. Έχω είπαμε ότι εγκρίθηκε. Η 197 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 108 ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 199 έχει αποσυρθεί και πάμε στη 200. Ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 30 το πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές έλεγχος τμήμα πρώτον της 30 είπαμε Πέρασε. Α, μικρή διαφορά. 28 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίθηκε με βραχία κεφαλή. Συνεχίζουμε στη 207, στη ίδια σελίδα κάτω-κάτω. Ψήφι υπέρ. 207. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 30, το δεύτερο τμήμα, ψηφιπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη 213 του κυρίου Ζέβερ, ψήφι Κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Διακόσια δεκαέξι, διακόσια δεκαεπτά, ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Η 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 35 υπέρ. Κατά. εγκρίνονται. Μήκος 20-19 Γκαρδίνη. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 220 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 221 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τσεκ. Ωραία. 221 ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρασε. 29 υπέρ 26 κατά. Εγκρίθηκε. Η 221 ήταν αυτή. Συνεχίζουμε. 222. Ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 223 ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 224 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 225 υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές ένοχος. Γιατί 225. Πέρασε. Mm. Απερίφθη. 25 υπέρ, 33 κατά. Κατά. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τσεκ. Καλά. Ελέγχουμε τη 226. Πέρασε. Το είχε απορριφθεί όμως. Σαφές. ...227 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας την ελέγξουμε αυτή. Παρακαλώ. Τη 227. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. 31 υπέρ, 26 κατά. Ευχαριστώ για το τσάι. Εγκρίνεται. Πάμε στη 232 υπέρ. 232 υπέρ. Κατά. Εποχές. απορρίπτεται. 233 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην επόμενη σελίδα. 245 είπε Κατά. 245 είπαμε. Ε, κατά. Κατά. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, έτσι. 244 και 246 μαζί ψήφι Κατά. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στη 18 σελίδα. Ε, η τροπολογία Γκαρντίνη, 246 ψήφι υπέρ, 64 συγγνώμη, 264 κατά. Αποχές απορρίπτεται. 265 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 268 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφτεται. Ορίστε. Κύριε Κράμερ. Έχετε λάθος στον κατάλογο της ψηφοφορίας σας. Εγώ είμαι εισηγητής. Στο 267 έχω βάλει θετικό πρόσημο, όχι αρνητικό. Μάλιστα. γιατί 267 ο εισηγητή είναι υπέρ. 267 Σνέλχαρτ Φλόρεντ. Ψήφι υπέρ τη τροπολογία αυτή. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42. 42. πίπτη λέει εδώ. 43 υπέρ. Κατά. Όχι. Απόχες εγκρίνεται, αλλά θέλετε να το ελέγξουμε. Για τη 43 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Und Abstimmung Πέρα στις ψηφορίες. Μικρή διαφορά, αλλά εγκρίθηκε. 28. Wo ε, είμαστε στη 271 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 272 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 273, 74, 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τσεκ. Καλά. Απερίφθη, με μία ψήφο διαφορά, αλλά απερίφθη, 28-29. 276. υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 44 και 277 είναι ίδιες, υπέρ. Κατά. Αποχές Έγκριντ. Τώρα, πού πάμε. Στι 45 και 278, υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Η ε, 279. Ψήφι πέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 279 θέλετε να την ελέγξουμε. Καλώς. Αρχίζει η ηλεκτρονική απορρίθευση για τη 279. Πέρας. 30 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίθηκε, αλλά κάπως εγώ τα καταλαβαίνω όταν εγκρίνονται. 280 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τσεκ. Για τη 49. Ηλεκτρονική επαλήθευση θέλετε. Καλά. Πέρας. Ε, πάντα οι ίδιες πλειοψηφίες είναι. 30 με 27. Οι συσχετισμοί είναι γνωστοί. 50. Ε, Υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Η 51 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Η 52 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Η 284 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. Και ερχόμαστε τώρα στην 285 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. 286 είπε. κατα Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 287-288 είπε. Ο Κράμερ θέλει έλεγχο. Πού, στη 286. Ναι. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Λοιπόν, 286 ζητάει ο κύριος Κράμερ, εισηγητής. Πέρας, ε, δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα, είχε εγκριθεί. Τι να κάνουμε τώρα. Ακόμα και αν ο εισηγητής ε, ε καταψηφίζει. 287-288, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Γυρνάμε σελίδα. 290. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 291-292 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 293 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δυστυχώς δεν φτάνει κυρίως και χάσατε. 295 ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Γιατί 295. Und beendet. Πέρασε. Ναι, 26 υπέρ, 30 κατά. Απορρίπτεται. 294 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 296 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 297-298 είναι οι ίδιες υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. 299 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 300 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 301 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 302 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 303 επέ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 304 επέ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 307. Συνεχίζουμε. επέ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 308 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 309. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 310 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 311 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 312 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 313 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 314 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 315 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τσεκ καλά τότε γιατί 315 ηλεκτρονική απολύθευση Πέρας. 25 υπέρ, 31 κατά, απορρίπτεται. 317 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 318 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 319 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 321 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 322 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 323 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 324 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 325 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 326 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 327 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 328 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 329 υπέρ. Έλεγχο για την 328 θέλετε. Καλά. Στο ΕΛΚ περισσεύει ένας. Βγάλτε κάποια κάρτα από το ΕΛΚ. Ε, τώρα εντάξει. Ε, πέρας 23 υπέρ 32 κατά, είναι σαφές κυρία Κλάς ότι έχει απορριφθεί. 329 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 330 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 3.31, 3.32 είναι οι ίδιες υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 3.33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.34 είπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 3.35 παρακαλώ. στις ψηφοφορίας. Ε, εγκρίθηκε αλλά με μικρή διαφορά. 338 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 339 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 340 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 341 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.43 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 346 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 347 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 348 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 348 θέλετε έλεγχο. Καλά. Ηλεκτρονική απολύθευση Ε, σαφέστερο δεν υπάρχει. 14. 1444. Ηλίου φαενότερ. 349. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 349. Μικρή διαφορά, όμως απερίφθη. 27 υπέρ, 29 κατά. 350-351 ίδιες, ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες, εγκρίνεται. 352 και 353 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μικρή διαφορά. Ε, νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Ας το ελέγξουμε. Δεν πειράζει. 3.52 και 3.53 μαζί. Πέρας. Α. Α, Λοιπόν, Πάμε τώρα σε αιτιολογικές σκέψεις. Recitals. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 57 και οι 55 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 58. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 58. 32 υπέρ, 26 κατά. Η 59 καταπίπτει και πάμε στην 60. Ψήφι υπέρ της 60. Κατά. Αφού έχεις έγκρινεται. Τσεκ. για την 60. Έλεγχος παρακαλώ. Α, τώρα δεν ψηφίζετε όλοι. Πέρασε. 32 υπέρ, 22 κατά, εγκρίθηκε. Ε, Αστιεύεσαι κρίση ή τα λες σοβαρά αυτά που λες. Το οποίο δεν ακούμε δυστυχώς. Λοιπόν, 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 1 υπέρ. Κατά. Αγωχέ. Έλεγχος. Για την τροπολογία παριθμόν 1, παρακαλώ. Πέρασε. 31-27 εγκρίνεται. Οι 2 και 64 μαζί ψήφι υπέρ. Κατά. ξέρω. 65. Είπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 είπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 είπε. Κατά. Αποχές. Απορρίφτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 72. Τσεκ. 71. Τσεκ. Abstimmung beendet. Ε, πέρας. Έχει υπορριφθεί. 26 υπέρ, 30 κατά. Ή 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφτεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 3 και 75 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4 τώρα ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ορίστε. Τεκ. Δεν με πιστεύετε, έλα. Ε? Τέσσερα. Η τροπολογία υπαριθμών 4. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Είναι σαφέστατο. 35 υπέρ, 23 κατά. 78 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται έτσι. Η οκτώ ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελειώσαμε. Θαυμάσια. Και ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, μία ψηφοφορία είναι. Αυτή. Δεν θα επαναληφθεί. Αρχίζει τώρα. Äh, Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται λοιπόν το νομοθετικό ψήφισμα 40 υπέρ 13 κατά και 4 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε εισηγητά Όλγκερ Κράμερ. Έχετε κάνει τρομακτική δουλειά. Μπράβο. Και όλοι οι σκιώδη εισηγητές αξίζουν Επένω και συγχαρητήρια καθώ επίση και η γραμματεία που ε, κατάφερε να κάνει αυτό το μεγάλο συμπίλημα για την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ είναι ε, μεγάλη νομοθετική δουλειά για το περιβάλλον αυτό που ψηφίσαμε και σε όγκο μεγάλη. Λοιπόν, έχουμε και άλλε ψηφοφορίε έτσι. Δεν τελειώσαμε. Είμαστε μέσα στα μέσα των ψηφοφοριών. Äh, ε, λοιπόν, το σημείο 9 στη μέση διάταξη. Και αυτό είναι καυτό θέμα. Δεύτερη ανάγνωση του Συμβουλίου για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ε, για τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλία και προϊόντα ξυλία στην αγορά. Η συγκίτρια είναι η κυρία Καρολάιν Λούκας, η οποία απουσιάζει και την αντικαθιστά η κυρία Σάτου Χάση. Δεν συζητάμε όμως, ψηφίζουμε. Έχουμε ενοποιημένες τροπολογίες. Δεν θέλετε να μας ακούσετε, αν δεν θέλετε δεν σας ενδιαφέρει, μήπως να βγείτε έξω για να μας διευκολύνετε, σας παρακαλώ. Όσοι συμμετέχετε στην ψηφοφορία, παρακαλώ να κάνετε τις συζητήσεις σας εκτός εθούσης. Έχουμε πολύ χώρο, έχουμε και καφενεία δίπλα. Ωραία. Έχουμε τις 8 τροπολογίες της πρώτης αυτές που λέει εδώ Consolidated Amendments. Η πρώτη ψήφι υπέρ, κατά, αβοχές εγκρίνεται. Δεύτερη, υπέρ, κατά άποχε εγκρίνεται 3 υπε. κατά άποχες εγκρίνεται Τέσσερα υπέ. κατά άποχες η πέντε, υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται η έξι. ορίστε η προφορική vote if there is no problem on voting on the... Ο κύριος Κυριακάκης, ε, έχω μια προφορική τροπολογία για την 6. Για το 6. Στην 117 έχω δικιά σας προφορική τροπολογία κύριε Σκυλακάκη, 117. An oral amendment on 6. Όχι, για την 6 έχω. €50,000 per annum. Äh, άρα αφορά την ε, ποιημένη έξι προφορική τροπολογία. Διαφωνεί κανείς να ψηφιστεί. Um, Κοιτάξτε, εξ ονόματος του εισηγητή που λείπει, της εισηγητρίας που λείπει, είμαι κατά της προφορικής τροπολογίας. Η εισηγήτρια θα την δεχόταν μόνον εάν ο συμβιβασμός, η συμβιβαστική δέσμη είχε αποτύχει. Εάν η αρχική 29 είχε απορριφθεί και εάν η εκτεταμένη χνηλασιμότητα, δηλαδή η 117, είχε εγκριθεί. Αλλά έχει ήδη απορριφθεί λόγω του συμβιβασμού, άρα είμαι κατά. Λοιπόν, υπάρχει αντίρρηση. Ήταν τόσο σημαντικό που σηκώθηκε και όρθια για να μιλήσει σαν του χάσει. Ναι. Λοιπόν, διαφωνεί κάποιο και δεν γίνεται δεκτή η προφορική τροπολογία και ψηφίζουμε την 6 αυτή την consolidated όπω είναι. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Υπέρ. Τη 7 τώρα. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ναι. Άρθρα ε, 19 υπέρ. Μετά. Απόχες. Εγκρίνεται. Έλεγχος για τη 19. Äh. Αρχίζει ψηφοφορία. Και τελειώνει τώρα. 32 υπέρ 24 κατά εγκρίνεται ναι. κυρία Βάισκερμπερ. Βεβαίω καταπίπτει 101 της Άνια Βάισκερμπερ και ερχόμαστε στην 21 και 23. Υπέρ τη 21 και τη 23. κατά Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Ναι. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Η 103 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 είπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τσεκ για την 24. ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει τώρα. Δουλεύουν τα μηχανήματα. 24 πέρας 31-24 εγκρίνεται σωστά τα είχα πει πάμε στην 105 ψήφι πέρα κατά αποχές απορρίπτεται 106 πέρα κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συνεχή. Στην 109 τώρα, έτσι. Υπέρ. Κατά. Ποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και μετά. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 της ηγήτριας υπέρ 8 Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Γυρνάμε σελίδα. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 30 υπέρ. άποχε εγκρίνεται. Η 31 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Η 119 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Η 120 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Η 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ο Λίζε θέλει έλεγχο. Εγώ σας λέω ότι εγκρίνεται. Για να δούμε την 32. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Δεν σας φτάσανε. 34-22. Ε, Με μεγάλη διαφορά εγκρίνεται κιόλας. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 124 υπέρ. 24 συγγνώμη. Κατά. Αποχές 35 υπέρ. αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 35. Παρακαλώ, αρχίζει τώρα. Äh, Κύριε Σνέρχαρτ, προηγουμένω περίσευε έτσι κι αλλιώ ένα του ΕΛΚΕ. Δεν χρειάστηκε να τρέχετε. Α, εντάξει, έβγαλε την κάρτα της κυρία Ζόμερ. Ωραία, ε, πέρας ψηφοφορίες. 23 υπέρ, 32 κατά. Ε, σαφέστατα έχει απορριφθεί. 125. 126. Έχει ε, αποσυρθεί 125. 126. Και αυτή έχει αποσυρθεί. Εντάξει. 128, 127 μαζί, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 38 είπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 133 είπε Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 134 είπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ξανάντα. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 42 με προφορική τροπολογία. Η του χάσει. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει πάλι να αντιταχθώ στην προφορική τροπολογία διότι αλλάζει τελείως την πρωτότυπη και αφαιρεί την κεντρική ιδέα της πρωτότυπης τροπολογίας και επιτρέπει στην Κομισιόν μόνο συμπληρώματα. Γι' αυτό είμαι κατά. Λοιπόν, ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο της 42. Υπέρ. Το αρχικό κείμενο, όχι την προφορική τροπολογία. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44-45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά Άποχες. Εγκρίνεται. Η 48 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 και 140 υπέρ και γυρίστε και σελίδα και 141 μαζί. Αυτές τις τρεις ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 142-143 είναι οι ίδιες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ορίστε. Η 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50, 150 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 επέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 πέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 57 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο. Ψήφι υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Ε, κατά.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 Und die ψηφοφορια ε, ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 24-30. 154 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχο θέλετε για την 67. Αφού είναι η ίδια πλειοψηφία πάντα. Έτσι, Έστω το ελέγξουμε, εν 67. Πέρασε. 29-27. Εγκρίνεται. 156 πέρα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το 58 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίψεις. 69 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 159 και 160 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 161-162 επίσης μαζί είπε. κατά αποχές εγκρίνονται 163-164 είπε. κατά 165-166 είπε. κατά αποχές εγκρίνονται 167 και 168 είπε. κατα κατά αποχές εγκρίνονται 169-170 υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε 70 και 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 172-173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Αιτιολογικές σκέψεις ακολουθούν τώρα. Η τροπολογία 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 73-74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Yeah. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 Υπέ. Αυτό είναι κατά, συγγνώμη. Αποχές απορρίφθηκε. Και τώρα, 77 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον, ψήφι Π. Του πρώτου τμήματο του 77. Κατά ποιο συγκρίνεται. Το δεύτερο ναι. υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83-84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 4 σε δύο τμήματα τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 5 υπέρ κατά Αποχές ε, εγκρίνεται. 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 93 κατευθείαν. Κάτω, κάτω στη σελίδα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίψετε. 11 υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεν κρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίψετε. Η 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 είπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 είπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 είπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψεται. 17 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και φτάσαμε αισίως στην τελική ψηφοφορία και εδώ. Είναι μία και μοναδική για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Αρχίζει τώρα ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρασε πω συντριπτική πλειοψηφία. 49 υπέρ, 6 κατά, δύο αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Καρολάιν Λούκας. Θα της θα πείτε κυρία Χάση και ε, σε όλους τους κοιόδης συγητές, στη γραμματεία. Έχετε κάνει τεράστια δουλειά όλοι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Και έτσι μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούμε να απαγορεύσουμε τις εισαγωγές λαθρέας ξυλίας, που έχει λατομηθεί λαθρέα δηλαδή. Äh, ε, συνεχίζουμε. Ε, την τρίτη μεγάλη ψηφοφορία έχουμε τώρα. Σχέδιο σύσταση σε δεύτερη ανάγνωση. Για τα νέα τρόφιμα. Η συγκίτρια είναι η κυρία Λιωτάρ. Δεν έχουμε ούτε συμβιβαστικές τροπολογίες, ούτε συλλογικές ενοποιημένε, αλλά πληθώρα με μονομένων τροπολογιών που πρέπει να ψηφίσουμε. Και αρχίζουμε από τη 38 της ηγήτρες. Ψήφι Π. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39. υπέ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40. Ε, ψηφοφορία κατά τμήματα. Τμήμα πρώτο. 4 τμήματα είναι. Αλλά όχι, τα ψηφίζουμε μαζί. Το πρώτο λοιπόν τμήμα κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 134, τμήμα πρώτο. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή, αλλά αν θέλετε συνελέγξουμε. Το δεύτερο τμήμα. Πέρασε. 29 υπέρ και 26 κατά εγκρίνεται και αυτή. Η 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. ε, συγγνώμη, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 50 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται η 51 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται η 52 είπε. κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στα δύο. Τσεκ θέλετε. Αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονική για τον έλεγχο της 61 παρακαλώ. Πέρασε. 15 υπέρ, 40 κατά, απορρίπτεται. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν εδώ. 62 υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 είπε. 100. Αποχές εγκρίνεται. 70 είπε. 100. Αποχές εγκρίνεται. 140 είπε. 100. Αποχές εγκρίνεται. 71 είπε. 100 αποχές εγκρίνεται. Η 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 73 στη σελίδα παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77. Με προφορική τροπολογία, ναι. παρακαλώ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ. Κατά. Okay. Ναι. Αποχές εγκρίνεται. 144 ναι. υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 86 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι εγκρίθηκε, αλλά το ελέξουμε για την 87. Πέρας.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 χωριστή ψηφοφορία, κατά τμήματα δηλαδή, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται τώρα αυτό. 95 υπέρ, κατά, αποχές, συγκρίνεται 96 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. άποχέ εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Τσεκ. Καλά. Ορίστε. Για την 100. Πέρασε. Α, μάλιστα. Απορρίπτεται λόγω Εκατόν 101. Ψήφι υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 102 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 103 είπε. κατά άποχες εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 χωριστή ψηφοφορία τμήμα πρώτο κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 ναι. υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 είπε, Κατά. Ε, εποχές εγκρίνεται. 111 είπε, Κατά. Έλεγχος με την 111 παρακαλώ. Πέρας. 11.31 ε, ε, υπέρ, 23 ε, κατά, εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 19 με προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 148. Ψήφι πέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 149 Υπέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 150 Υπέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 είπε. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 117 είπε. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 118 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 119 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 120 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 121 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 124 είπε. 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 3 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ή 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ή 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η εννέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δέκα. χωρίς την ψηφοφορία τμήμα πρώτο ΦΥΠΕ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ κατά Έλεγχος χρειάζεται εδώ. Για το δεύτερο τμήμα της 10. Ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ. Πέρας. και αν χρειαζότανε. 28 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 11 υπέρ.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 Πέρας. Πέρας. Μα σαφέστατο ήτανε. Σαφέστατο. Αγαπητέ συνάδελφοι, κύριε Ρώση. Η 18 ήταν αυτή, πάει απορρίφθη, 19. υπέ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 είπε. Κατά. Α. Αποχές. Απορρίπτεται. Ναι. 21 είπε. κατά άποχες εγκρίνεται 22 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 23 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 24 υπέρ κατά από άποχες απορρίπτεται 128 υπέρ κατά Ε, νομίζω ότι είχε απορριφθεί. Α το ελέγξουμε όμως. 128. Abstimmung jetzt dann beendet. Πέρασε. Ναι. Απερίφθη. 25. Πέρα. Κατά αποχές απορρίπτεται 26 Είπε; κατά αποχές απορρίπτεται 129 Είπε; κατά αποχές εγκρίνεται 28 Είπε; κατά αποχές εγκρίνεται. 29 είπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ή 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ή 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά έλεγχος παρακαλώ για την 33 ε, πέρας ε, της ψηφοφορίας 29 υπέρ 25 κατά. Εγκρίθηκε. Οι Η 34 ψήφι υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφτεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. Και η 133 με προφορική ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Δουλέψαμε θαυμάσια και φτάσαμε στην τελική ψηφοφορία που είναι μία και μοναδική, αρχίζει τώρα, για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Πέρασε. 49 υπέρ, 2 κατά, 3 αποχές, συγχαρητήρια κυρία Λιωτάρ. Συγχαρητήρια και σε όλους τους κοιόδης ηγητές και τη γραμματεία για το έργο τους. Δουλέψαμε καλά σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Ήταν πολλέ οι ψηφοφορίες, εκατοντάδε οι τροπολογίε. Ο Επίτροπος κύριο Ντάλι αυτή τη στιγμή είναι στην Επιτροπή Γεωργίας και θα έρθει όπω έχει προγραμματιστεί στι 11 και 4. Τώρα έχουμε μισή ώρα διάλειμμα, το οποίο αξίζουμε όμω. Ε, και τέταρτο, ελάτε όμως ακριβώς την ώρα σας για να δούμε τον Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ. Διακοπή, μικρό διάλειμμα.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 Μιλήσαμε για την προστασία του περιβάλλοντος και θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο και τους συνεργάτες του, ο οποίος θα αναφερθεί σε θέματα υγείας. Εμείς ακούσαμε <clears throat> την τελευταία φορά τον κύριο Επίτροπο στα πλαίσια της ακροάσεως που είχαμε οργανώσει για τα θέματα που άπτονται της υγείας. Τώρα προσπαθούμε να καθορίσουμε το νέο πρόγραμμα εργασίας, θα έλεγα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα αρμόδια κομμάτια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ακούσουμε κύριε Επίτροπε την παρουσίασή σας και μετά θα περάσουμε στην διαδικασία των ερωτήσεων. Δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο στον κύριο Ντάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόλις ήρθα από την Επιτροπή Γεωργίας και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Πρόεδρε, αγαπητοί μέλη, είναι μεγάλη χαρά που είμαι μπροστά σας για πρώτη φορά μετά από την ακρόασή μου τον προηγούμενο Ιανουάριο. Έχει μεγάλη σημασία να δείξω ότι είμαι αποφασισμένος να είμαι σε στενό διάλογο με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι πεπισμένος ότι παίζεται ένα κρίσιμο ρόλο και οι εργασίες των θεσμικών οργάνων πάντα στοχεύουν την αποτελεσματικότητα, στην αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Στο εφόμενο στο πρόγραμμα της Επιτροπής για το 2010 να σας περιγράψω το πλαίσιο για τις προτεραιότητες τις οποίες θα επιδιώξουμε και θα κινηθούμε. Η Ευρώπη 2020, το πρόγραμμα αυτό, είναι ε, θα έλεγα ένα πρόγραμμα για μορφές ανάπτυξης αηφόρες και συστηματικές. Ο τομέας για τον οποίο είμαστε υπεύθυνοι έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει για να προωθήσει αυτές τις ε, προσπάθειες είτε μέσω της βελτίωσης της υγείας είτε μέσω της ε, ε, φροντίδας της αλυσίδας της τροφιμικής και των καινοτομιών γενικότερα που θα πρέπει να βοηθήσουν τους καταναλωτές να κάνουν σωστές επιλογές. Πέρυσι είχαμε την πανδημία της γρήπης ήταν θα έλεγα ένα ουσιαστικό παράδειγμα αντιμετώπισης μιας κρίσης και σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα μαθήματα στα οποία καταλήξαμε από την εμπειρία αυτή, να βελτιώσουμε και να ρυθμίσουμε σωστά το σύστημά μας έτσι ώστε να είναι πιο σωστά προπαρασκευασμένο την επόμενη φορά. Χαίρομαι για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις προσπάθειες αυτές, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε πιθανές μελλοντικές ε, πανδημίες. Τον Φεβρουάριο σας ζητήσαμε να στείλετε εκπροσώπους εφόσον το επιθυμείτε για τη διαδικασία αξιολόγησης. Σας έστειλα και μία πρώτη αξιολόγηση των τεσσάρων πρώτων μηνών της πανδημίας και μετά από λίγους μήνες θα σας στείλω επίσης και στοιχεία για τη χορήγηση των εμβολίων κτλ. σε διεθνές επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε μέρος ε, στην ε, επανεξέταση των κανονισμών στον τομέα των πανδημιών από την Διεθνή Οργάνωση, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Συνεργαστήκαμε με τον Παγκόσμιο αυτό οργανισμό και για τον καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών προπαρασκευής ε, για την αντιμετώπιση των πανδημιών Όλα αυτά θα φανούν και στην τελική πρόταση την οποία θα κάνουμε στο τέλος του χρόνου έτσι ώστε ε, να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε σωστά τέτοιες εκδηλώσεις πανδημίας και γρήπης ε, στο μέλλον. Για το καπνό. Ξέρουμε ότι ο καπνός ε, σκοτώνει, ξέρουμε ότι ο καπνός κάνει εξαρτημένα τα άτομα που τον χρησιμοποιούν και υποφέρουμε γενικότερα από τη χρήση του. Και γι' αυτό θα καταθέσω μία πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας παραγωγής καπνού. Ε, υπάρχουν νέα προϊόντα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που προκαλεί ο καπνός και να προστατεύσουμε τους νέους. Κατά τη διάρκεια της εντολής μου θέλω επίσης να ε, μεταρρυθμίσουμε τις οδηγίες για για τον έλεγχο των ιατρικών προϊόντων και των φαρμάκων τα οποία χρησιμοποιούνται για τα θέματα αυτά. Είναι πρωτοβουλίες χρήσιμες και για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και για την απομάκρυνση των γραφειοκρατικών εμποδίων και για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στην αναθεώρηση της οδηγίας για τα ιατρικά εργαλεία όπως επίσης και για τις διαγνώσεις in vitro Θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους καταναλωτές και ασθενείς στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα του τομέα αυτού δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν. Να στραφώ τώρα σε κάποια ευαίσθητα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν και εσάς και εμένα με τον ίδιο τρόπο. Ξεκινάω με, τις, με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ας ξεχωρίσω την αδειοδότηση με την καλλιέργεια. Η βασική μου αντίληψη είναι απλή. Δεν είμαι υπέρ, δεν είμαι κατά των γενετικά τροποποιημένων. Ακολουθώ όμως τις λήψεις αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο επιστημονικής τεκμηρίωσης. Όταν μια επιστημονική ομάδα θεωρεί ότι καλύπτονται κάποιες ε, νομικές εν προϋποθέσεις, δεν θα κολλησιεργήσω εγώ για την αδειοδότηση. Και δεν θα πρέπει εμείς ε, να θεωρηθούμε οπισθοφυλακοί στον τομέα των καινοτομιών. Σε επίπεδο αδειοδοτήσεων, οι διαδικασίες που αποφασίστηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2003 παραμένουν το σημείο εκκίνησης. Πρέπει να είναι ψύχρεμη η συζήτηση για τους γενετικά τροποποιημένους μηχανισμούς και προϊόντα. Πρέπει να γίνει σε ορθολογικό επίπεδο. Έχω πει σε όλους τους εταίρους ότι θα πρέπει να υπάρξει σωστή ενημέρωση για τα γενετικά τροποποιημένα. Θα πρέπει επίσης να μην υπάρχουν στην παραγωγή γενετικά στοιχεία τα οποία να προκαλούν προβλήματα και θα πρέπει ταυτόχρονα να μπορούμε να παρακολουθήσουμε με συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο τρόπο την καλλιέργεια των γενετικών τροποποιημένων έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε σωστά τα υπέρ και τα κατά. Την επόμενη Πέμπτη θα συζητήσω τα θέματα αυτά με όσους εμπλέκονται για να εξετάσω τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους. Σχετικά με την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων, ξέρετε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Επιτροπή πριν το καλοκαίρι με μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για το πώς θα δώσουμε την δυνατότητα στα κράτη να αφήσουν ή να μην αφήσουν την κυκλοφορία στο έδαφος τους των συγκεκριμένων αυτών ε, προϊόντων. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία την χάνει πλήρως της υποστήριξής μου και καλύπτεται επίσης και από τις κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου Μπαρόζου, ε, οι οποίες έχουν ήδη ε, κυκλοφορήσει. Για την κλωνοποίηση τώρα. Τον Φεβρουάριο είχα πει ότι θα προετοιμάσω μια έκθεση μέχρι το τέλος του χρόνου και ε, αυτό είναι κομμάτι του προγράμματος εργασίας. Θέλω να ετοιμάσω μια αντίληψη ε, ολοκληρωμένη σε σχέση με την κλωνοποίηση. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι σε επαφή με όλους τους εμπλεκομένους έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια εξισορροπημένη άποψη. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσά θα ενδιαφερθείτε γι' αυτό. Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει επίσης την αναθεώρηση της χρηματοδότησης των συστημάτων ελέγχου για τα τρόφιμα και την τροφιμική αλυσίδα. Νομίζω ότι αυτό θα βασιστεί στην αντίστοιχη προσπάθεια που ξεκινήσαμε το 2008. Η αναθεώρηση αυτή έχει σαν στόχο την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων ε, σχετικά και με το τίμημα των ελέγχων, έτσι ώστε τα κράτη να έχουν περισσότερα μέσα οικονομικά στη διάθεσή τους και να εξετάσουμε επίσης ε, και το θέμα της εμπορίας της σπορίας έτσι ώστε ε, να μην εξαιρείται ουσιαστικά η σπορία από ό,τι ισχύει για την εσωτερική αγορά. Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει τις εξής προτεραιότητες. Μια νέα νομοθετική ρύθμιση για την υγεία και ευημερία των ζώων, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την ευημερία των ζώων. Ε, όπως επίσης υπάρχει και νέα προσπάθεια για τον κανονισμό για τη μεταφορά των ζώων και αυτό δείχνει τι βάρος δίνουμε στον συγκεκριμένο τομέα. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το πρόγραμμα εργασίας για το 2010 και πέραν του 2010 θα πρέπει να είναι καινοτομικό να σας πω τι εννοώ προς την κατεύθυνση της επιστημονικής πρόοδου. Είμαι υπέρ της καινοτομίας και θέλω να μεγιστοποιήσω τα πλεονεκτήματα τα οποία μπορεί να μας δώσει η καινοτομία αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Είμαι υπέρ της υπεύθυνη της έλογης καινοτομία σεβόμενοι τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν σε επίπεδο κινδύνων και ασφάλειας μπορούμε να εξηγήσουμε και πρέπει να εξηγήσουμε τα προϊόντα στους καταναλωτές. Η εμπιστοσύνη δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη και δεν θα πρέπει να οδηγούμεθα σε καταστάσεις από πλευράς της βιομηχανίας η οποία προσπαθεί να μονοπολίσει την ενημέρωση προς την κοινωνία και να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων. Απαιτείται σε σχέση με την επιστήμη μια ξεκάθαρα ανοιχτή συζήτηση στην οποία να συμμετέχει και η βιομηχανία που αναπτύσσει νέα προϊόντα και νέες διαδικασίες έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τους φόβους και τις επιφυλάξεις. Νομίζω ότι θα με υποστηρίξετε και προς την κατεύθυνση αυτή προχωρώντας τη συζήτηση γύρω και από το θέμα της ασφαλείας των τροφίμων. Τώρα να να ασχοληθώ με κάποια θέματα που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο παρελθόν στο πρόγραμμα εργασίας για τις φαρμακευτικές ουσίες. Έχει υπάρξει εξαιρετικό αποτέλεσμα στις διοργανικές διαπραγματεύσεις και ελπίζω αυτό ε, να ισχύσει και για το κομμάτι που θα αφορά την ενημέρωση προς τους ασθενείς. Απαιτείται να υπάρξει αυτό. Πρέπει να υπάρξει σωστή ενημέρωση για ιατρικά προϊόντα. Και αυτό ισχύει σε πιο πολλές χώρες ανεξάρτητα της νομοθετικής ή μη ρύθμισης του θέματος. Η γνώση είναι το καλύτερο μέσο που μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες μας. Θα πρέπει οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικού επίπεδου πληροφορίες, ποιοτικέ πληροφορίες. Αυτή είναι η στόχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους ασθενείς να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες να είναι ενήμερες των, του ωφέλους και των προβλημάτων που μπορεί να υπάρξουν. Αυτή τη στιγμή έχει ψηφίσει το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Θα εξετάσω τις τροπολογίες σας και από πλευράς ασθενών θα έλεγα. Ε, για τις διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας. Θα ήθελα να πω ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας ανεπίσημης του Συμβουλίου Υπουργών Υγείας η Ισπανική Προεδρία έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Είμαι αισιόδοξο για την προοπτική μια συμφωνίας η οποία θα πρέπει να καταλήξει στο Συμβούλιο ίσως και τον μήνα Ιούνιο το Συμβούλιο και το κείμενο του Συμβουλίου ίσως να μην είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα επιθυμούσαμε. Παρ' όλα αυτά όμως μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση τώρα έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να πάρει τις αποφάσεις του όταν αυτό πρέπει το ταχύτερο δυνατόν σε δεύτερη ανάγνωση. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα προσφύγουμε για μια ακόμη φορά σε εσά όταν έχουμε ανάγκη. Σχετικά τώρα για τις αναφορές και τα παράπονα σε σχέση με τα τρόφιμα. Βλέπουμε ποιες είναι οι ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις αναφορές αυτές σταδιακά σχετικά με τις ουσίες και ε, το περιεχόμενο και την ενημέρωση για το περιεχόμενο προϊόντων ιδιαίτερα προϊόντων τα οποία περιλαμβάνουν υψηλά επίπεδα λίπους, άλατος ή ε, ζάχαρης. Πράγματι ορισμένα τέτοια προϊόντα δεν μπορεί να διαφημίζονται σαν επωφελή για την υγεία των καταναλωτών. Και γι' αυτό το ε, Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει μια τροπολογία στο παρελθόν που αναιρεί αυτή την δυνατότητα. Πάντως αυτά τα τροφιμικά προφίλ τα οποία περιλαμβάνονται μερικές φορές στα προϊόντα όταν κυκλοφορούν βοηθούν τους καταναλωτές να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, νομίζω ότι σας παρουσίασα συνοπτικά και γρήγορα τους ε, βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις τελευταίες εξελίξεις. Το πρόγραμμα εργασίας δεν αντικατοπτρίζει το σύνολο των θεμάτων που θα ήθελαν ορισμένοι. Και νομίζω ότι ο οδικός χάρτης που θα ακολουθήσει και οι προτάσεις μας στο μέλλον θα είναι να κάνουμε προτάσει για μια σύγχρονη αντιμετώπιση ε, των προβλημάτων της υγείας μετά το 2011. Είμαι στη διάθεσή σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε Τζον Ντάλι για την παρουσίαση των θεμάτων σας, των αρμοδιοτήτων και τις τάσεις που θέλετε να ακολουθήσετε στις αποφάσεις σας. Το περιβάλλον είναι καυτό το θέμα βέβαια, αλλά ακόμα πιο ευαίσθητο και καυτό είναι το θέμα της δημόσιας υγείας στην κοινή γνώμη και αναφερθήκατε και σε θέματα που απασχολούν ε, πολλοί του πολίτες. Πάνω από 20 συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Σας παρακαλώ αυστηρά δίλεπτο έκαστος, Αλλιώ αυτό είναι άδικο απέναντι στους άλλου συναδέλφου. Αρχίζουμε αμέσως. Κλείνω και τον κατάλογο μιλητών, έτσι. 20 φτάνει και παραφτάνει. Από το Λαϊκό Κόμμα, ο Ρίχαρτ που παίρνει τηλέφωνο του, <laughs> αλλά Λίζε, εν πάση περιπτώσει. Δύο λεπτά και το ρολόι αρχίζει τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Βεβαίω ε, είστε δικαιολογημένο για την καθυστέρηση. Ε, εφόσον ήσασταν σε άλλο όργανο του Κοινοβουλίου. Αλλιώ, αν είχατε άλλη δικαιολογία, δεν θα τη δεχόμασταν. Έχω τις εξή παρατηρήσεις. Στην ε, ακρόασή σας μας είχατε πει για τις οργανώσεις ε, των ασθενών που θέλετε στο μέλλον να τις υποστηρίξετε ε, περισσότερο και μάλιστα τις ανεξάρτητες ενώσεις των ασθενών. Έχετε συγκεκριμένες σκέψεις να μοιραστείτε σήμερα μαζί μας. Δεύτερον, αναφερθήκατε στην κλωνοποίηση. Ε, μόλις ψηφίσαμε για την έκθεση Λιωτάρ για τον κανονισμό για τα νέα τρόφιμα, Novel Food και ξέρουμε ότι θέλετε ξεχωριστή πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς ε, ζητούμε και απαγόρευση μάλιστα. Ε, παρακαλώ να επιταχύνετε πολύ τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλιώς θα συγκρουστούμε με τον κανονισμό Novel Food αν δεν κάνει καθόλου πρόταση η Κομισιόν. Το δικαίωμα πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίω και θα πρέπει να γίνει σεβαστό, αλλά αν θέλετε να περάσει γρήγορα αυτή η υπόθεση Novel Food, χρειαζόμαστε χωριστή πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα ε, γρήγορα. Μιλήσατε για τον καπνό τελευταίο. Σωστό το θεωρώ αυτό που λέτε για τα προϊόντα καπνού και τη σχετική οδηγία να σκεφτούμε πώ μπορούμε να προστατεύσουμε ακόμα καλύτερα τον κόσμο. Θα σα παρακαλούσα να διευκρινίσετε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι Δεν θα έχουμε πανευρωπαϊκά ε, απαγόρευση ε, καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Ο κόσμος είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα της επικουρικότητας και μπορεί να μας γίνει μπούμεραν αυτή η υπόθεση. Ας απαγορεύουν τα κράτη ξεχωριστά που επιτρέπεται το κάπνισμα και που όχι. Όχι μια πανευρωπαϊκή ρύθμιση. Και θα, ε, παρακαλώ να δεσμευτείτε και για την απαγόρευση ενισχύσεων στους καπνοπαραγωγούς στην καλλιέργεια. Ε, η Σας κατευχαριστώ. Δεν το είπατε τελείως ακριβώς το όνομά μου, αλλά πάντων ευχαριστώ κύριε Ντάλι. Έχω ασχοληθεί πολλές φορές με τον καπνό και μου άρεσαν αυτά που είπατε για αυτόν. Αλλά εμεί περιμέναμε τέσσερα χρόνια η Κομισιόν να μας ε, εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτά τα... Ε, αυτές οι θρεπτικές αναλύσεις που να περιλαμβάνουν και τα λίπη και τη ζάχαρη και οι οργανώσεις των καταναλωτών είναι αμφίβολο αν σε αυτή την περίπτωση θα επέτρεπαν τα ντόνατς και ε, άλλα διάφορα είδη μπισκότων που έχουν πολύ ζάχαρη. Η Κομισιόν λοιπόν πρέπει να διασφαλίσει ότι θα πετύχουμε ακριβώς τους στόχους που επανειλημμένα έχουμε ζητήσει. Στον πολύ Κορίν Λεπάζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την προσέλευσή σας. Έχω δύο ερωτήματα για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Μας μιλήσατε για εθνικοποίηση στην οποία επιμένει ο πρόεδρος Μπαρόσο. Αλλά σε συνδυασμό με τα αιτήματα του Συμβουλίου Υπουργών του περασμένου Δεκεμβρίου που ζήτησε ανατίμηση, επανεξέταση των τρόπων ανάλυσης, τι θα κάνετε. Και εδώ έρχεται το δεύτερο μου ερώτημα, δηλαδή θέλετε να υποβάλλετε καμία πρόταση για αυτό το θέμα που είναι ουσιώδες και είναι θέμα επιστημονικής, αντικειμενικής αξιολόγησης μετά από διαβούλευση βέβαια με εμπειρογνώμονες εφόσον βέβαια η εμπιστοσύνη που θα έχουμε στους εμπειρογνώμονες αυτούς είναι εγγυημένη και εφόσον υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής ερωτώ πώς τι θα κάνετε, θα συνδεθεί το Κοινοβούλιο με την ανάλυση αυτή, θα προτείνετε τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας και τις επιλογές της ΦΣΑ ή ΕΦΣΑ ώστε η υγεία των καταναλωτών και καταναλωτριών να μπορεί να τύχει κάποια εγγύηση για να έχουν κάποια εμπιστοσύνη οι καταναλωτές και οι καταναλώτριες για τις αποφάσεις που παίρνει η Ένωση. Ευχαριστούμε. Μισελ Ρεβάζη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω τον κύριο Ντάλι. Δύο ερωτήματα. Είχατε πει για την παρασμένη γρήπη ότι θέλετε να πάρετε μαθήματα. Λοιπόν, εμείς οι βουλευτές και εμείς θέλουμε να κάνουμε τον έλεγχό μας και ζητούμε μια προσωρινή επιτροπή. Έχουμε 210 υπογραφές. Ελπίζω οι βουλευτές και ο Επίτροπος να συμφωνούν γι' αυτό. Αλλά θέλω και εγώ να ρωτήσω κάτι για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Εγώ εξεπλάγει είμαι βιολόγος, επιστήμων και ξέρω ότι στις καινούργιες πατάτες υπάρχει ένα πολύ ανθεκτικό γονίδιο στην ε, ένα είδος αντιβιωτικού το οποίο νεομικίνη, ένα είδος νεομικίνης και με εξέπληξε το ότι όταν το εγκρίνατε δεχτήκατε την ύπαρξη αυτού του γονιδίου στην πατάτα και είπατε ότι θα είναι μόνο για τη διατροφή των ζώων. Αλλά τελικά αυτό δεν αποκλεί και να περάσει και στην ε, ανθρώπινη διατροφή σε μια τάξη 0,9% είναι η νομική αυτή κατά της φυματίωσης. Θα ήθελα λοιπόν να μου δικαιολογήσετε γιατί δεχτήκατε αυτή τη γενετικό τροποποιημένη πατάτα. Η κυρία Καρτή Καλιοτάρ και μετά Επίτροπος να απαντήσει, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι πάρα πολύ που μας είπατε ότι ε, η πολιτική τροφίμων θα πρέπει να βελτιωθεί και να είναι καλύτερη για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά έχω μια ερωτησούλα να σας κάνω. Μ' ακούτε κύριε Ντάλη ή συζητάτε. Α, εντάξει, ευχαριστώ. Ε, μπορείτε να διαψεύσετε ότι ήδη έχετε αρχίσει διαπραγματεύσει ή πρόκειται να συμφωνήσετε με τις Ηνωμένε Πολιτείε για άλλες ιδέες ε, νομοθεσίας για ε, την κλωνοποίηση και για τα ζώα τα κλωνοποιημένα και ποια είναι η στρατηγική σας ε, χωρίς να μας έχετε δώσει ακόμα επίσημη θέση και στο Κοινοβούλιο μόλις ακούστηκαν μεγάλες επιφυλάξεις. Στην πλειοψηφία του το Κοινοβούλιο ζήτησε ε, ότι θέλει ρύθμιση που να πηγαίνει στην κατεύθυνση απαγόρευσης. Λοιπόν, διαψεύδεται ότι έχετε αρχίσει διαπραγματεύσεις, γιατί ε, έχω πάρει εγώ διάφορα ανώνυμα email. Αυτά είναι πλαστά. Ε, ποια είναι λοιπόν η θέση σας και πρώτα να διαμορφώσετε θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά να πάτε σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Äh, Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Ε, απαντήστε κύριε Επίτροπε, παρακαλώ. Για τις οργανώσεις των ασθενών, κατά την ακρόαση μου είχα πει ότι θα εξετάσω την περίπτωση να δεχτώ ορισμένε νέες δυνατότητες χρηματοδότησης αυτών των οργανώσεων καταναλωτών, καταναλωτριών και ασθενών που είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Προς στιγμήν ακόμη το σκεφτόμαστε και το μελετάμε τη δυνατότητα δηλαδή αυτήν και θα καταλήξουμε σε κάποιου είδους προτάσεις για να τις συζητήσετε μαζί μας. Ελπίζω, ελπίζω σύντομα. Για την κλωνοποίηση είχαμε πει, είχαμε υποσχεθεί ότι στο τέλος του χρόνου θα κάνουμε μια έκθεση και θα το πράξουμε. Δεν ξέρω όμως τι ηλεκτρονική βασικό μήνυμα είναι αυτό που αναφέρατε κυρία Λεωτάρ. Δεν το ξέρω. Μπορώ όμως να σας πω με τα βεβαιότητος ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες ή με οποιονδήποτε άλλον ως προς την κλωνοποίηση. Θα πραγματοποιήσουμε διαλόγους ήδη τους πραγματοποιούμε με όλους τους ενδιαφερόμενους και τις Ηνωμένε Πολιτείες και άλλους. Τις έχουμε καλέσει και αυτές σε διάλογο αλλά δεν έχει αρχίσει καμία διαπραγμάτευση. Ούτε σχεδιάζεται καμία ακόμη γιατί πρέπει πρώτα η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει κάποια πολιτική και μετά να την υποστηρίξει σε διαπραγματεύσεις. Για τον Καπινό και το αν θα υπάρξει πανενοσιακή απαγόρευσή τους, του καπνίσματος, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να επιμείνω να υπάρξει νομοθεσία σχετικώς, αλλά θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με τις απαγορεύσεις που έχουμε ήδη ζητήσει. Από ό,τι γνωρίζω οι επιχορηγήσεις για τα προϊόντα καπινού έχουν καταργηθεί. Θα καταργηθούν από του χρόνου μάλλον. Και αυτό δημιουργεί βέβαια πρόβλημα διότι όπως όλοι γνωρίζετε η χρηματοδότηση για την αντικαπνιστική εκστρατεία από αυτό το ταμείο το Γεωργικό Ταμείο προέρχεται και τώρα δεν υπάρχει πια αυτό το ταμείο, δεν υπάρχουν χρήματα και ελπίζω με τη βοήθειά σας να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε την αντικαπινιστική εκστρατεία. Για τις τροφιμικές αναλύσεις Είχε υποθεί ότι βάλαμε πολύ ψηλά όρια, ανώτατα όρια. Αλλά βασιστήκαμε σε επιστημονικά δεδομένα. Δεν το κάναμε αυθαίρετα. Έχουμε ένα σύστημα γνωμοδοτήσεων και από την άλλη, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, σημείωσα ότι η Επιτροπή σας δεν δέχεται στους, νέες, ε, στους νέους διακανονισμούς για τα τρόφιμα να υπάρχει αυτή η συστηματική ανάλυση. Αυτό θα ζητήσω να αλλάχθεί διότι κατ' εμάς τα ε, στοιχεία για τη διατροφή είναι πολύ σημαντικά. Γιατί τι λέμε εμείς, ότι όλα, κάθε προϊόν που επιτρέπεται να διατεθεί στην αγορά ως ωφέλιμο για τον καταναλωτή και την καταναλώτρια για οποιοδήποτε λόγο δεν θα έχει το δικαίωμα να το πράξει με αυτή τη διαφήμιση αν δεν αναφέρει επίσης ποια είναι τα ποσοστά των τροφιμικών ουσιών που περιέχει. Διότι αν δεν πληροφορούμε τον καταναλωτή και την καταναλώτρια για τα στοιχεία αυτά, τότε νομίζω ότι δεν θα τον εξυπηρετούμε ή δεν θα την εξυπηρετούμε. Και έτσι νομίζω θα αυξάναμε τη δυνατότητα εξαπάτησης για τα γενετικώς τροποποιημένα. Και στην Επιτροπή Γεώρ Άγκρη μου θέσανε πολλά τέτοια ερωτήματα και είχα πει ότι το θέμα αυτό πρέπει να το συζητήσουμε όσο δυνατόν επιστημονικότερα. Ένας βουλευτής μάλιστα είπε μήπως δεν θα μπορούσαν από κοινού οι Γεώρ και οι Περίβ να συνεδριάσουν και να το συζητήσουν. Και εγώ είμαι υπέρ μια συζήτησης τόσο ανοιχτής ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα, ποιες είναι οι επιπτώσεις των αποφάσεών μας και οι εμπειρογνώμονες μας λένε μέχρι τώρα ότι οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί που έχουν εγκριθεί είναι ασφαλείς. Και εμείς ως Κομισιόν το μόνο που μπορούμε να κάνουμε που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε με απόφαση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου είναι να εφαρμόσουμε αυτά που μας λένε οι επιστημονικές αναλύσεις. Εγώ δεν μπορώ ως επίτροπος να αυθαίρετα να πάρω με αποφάσεις για το τι μπορεί να εγκριθεί και τι δεν μπορεί. Και αυτό είναι σωστό και πρέπει. Πρέπει να είμαι ουδέτερος και αντικειμενικός. Να στηρίζομαι δηλαδή στην επιστημονική συμβουλή που θα μου έχουν δώσει. Αυτό κάναμε. Not... Όσο για το γονίδιο εκείνο που είναι αντιφηματικό, δεν ξέρω τίποτα. Είναι βιομηχανικό προϊόν και βιομηχανικό θα παραμείνει, όχι διατροφής. Το αντιφηματικό γονίδιο έχει αναλυθεί και συζητηθεί και εκτιμηθεί όχι μόνο από την ΕΦΣΑ αλλά και από την ECDC και την ΜΕΑ για να κάνουν και αυτές τις εκτιμήσεις τους και να δουν κατά πόσον είναι ασφαλές και τελικά κατέληξαν όλοι ότι είναι ασφαλές. Για τη γρήπη ή τα 1 1 όπως είπα ακόμη κάνουμε τη μελέτη και καλέσαμε και την Επιτροπή σας να συμμετάσχει στην αποτίμησή μας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε γιατί θέλω να σας τονίσω ένα πράγμα οι πανδημίες θα ξαναγίνουν, θα ξανασυμβούν και φοβάμαι Φοβάμαι λέγω ότι ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστούμε αυτή τη φορά την πανδημία μπορεί να δημιουργήσει το σύνδρομο του λύκου και για τα θεσμικά όργανα και για τις χώρες μέλη. Δηλαδή να θεωρηθεί ότι είμαστε υπερβολικοί και ότι τελικά μπορούμε να σταυρώσουμε τα χέρια, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα και έτσι να μην αντιδράσουμε όπως θα έπρεπε και να διακινδυνεύσουμε τη ζωή των πολιτών μας. Ευχαριστούμε πολύ για τα τροποποιημένα. Υπήρξαν επαφές μεταξύ μου και του Προέδρου της ΓΕΟΡ και εξετάζουμε όντως την περίπτωση να κάνουμε μια κοινή συνεδρίαση. Πρέπει όμως να είστε λίγο συντομότερος γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ακούγοντάς σας βλέπω πόσο τεράστια είναι τα... τεράστιες είναι οι ευθύνες σας για τις διαμεθοριακές οδηγίες ως προς τα θέματα υγείας. Η Ισπανική Προεδρία είπε ότι έχει τη θέληση να κάνει κάτι και μέχρι τις 8 Μαΐου έπρεπε τα κράτη-μέλη να δηλώσουν τις θέσεις τους. Υπήρχε ακόμη το πρόβλημα του, των ορισμών, παραδείγματο χάρη του προβλήματος των Βρετανών ε, που είχαν πάρει τη σύνταξή τους στην Ισπανία και αν πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις ακόμη και αν υπάρχει πρόβλημα ποιότητας της υγείας, το θέμα της ήττα υγείας. Γι' αυτό κύριε Επίτροπε θα ήθελα να μου πείτε τι συμβαίνει με όλα αυτά για να μπορέσουμε και εμείς να το αποφασίσουμε σε δεύτερη ανάγνωση. Τέλος, για τα πλαστά φάρμακα ή νομίζω ότι δεν είχαμε υπάρξει αρκετά απαιτητικοί διότι δεχτήκαμε τη δυνατότητα του repackaging. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποια ρήτρα που να διασφαλίζει περισσότερη ασφάλεια εφόσον δεχόμαστε το repackaging. Μπορείτε να μας δώσετε καμία πρόσθετη εγγύηση. Ευχαριστούμε Τζίλες. Σίλτερς δηλαδή. Και εγώ για τη δημόσια υγεία. Η Ένωση άρχισε να εφαρμόζει ένα κοινό πρόγραμμα έρευνας για τα τρόφιμα για καλύτερο συντονισμό ορισμένων βαφών Θα έπρεπε όμως να γίνει κάποια μεγαλύτερη προσπάθεια και για τις επιπτώσεις καταναλώσεως συνοπνεύματος που είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παράγοντας δημιουργίας χρονίων παθήσεων στον κόσμο. Τα συμπεράσματα της Σουηδικής Προεδρίας ζητούσαν κάτι πιο τολμηρό, όπως αυστηρότερες υψηλότερες τιμές. Ευχαριστούμε, Ρενάτα Ζάμερ. Η κυρία Ζόμερ, ευχαριστώ. Χαίρομαι που σας βλέπω κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να επανέλθω στα θέματα των προφίλ διατροφικής ε, ηθροπτικής αξίας. Ξέρετε ότι έχει απορριφθεί για δεύτερη φορά αυτή η πρόταση. Να σας πω γιατί. Διότι αυτά τα προφίλ της διατροφικής αξίας ακριβώς δεν έχουν αξία. Δεν έχουν πραγματική τεκμηρίωση και επιστημονική ε, βάση. Παρ' όλα αυτά το χρησιμοποιείται ως βάση και ε, για την εγκυρότητα των ε, ισχυρισμών υγείας, των λεγόμενων health claims. Και βέβαια θα πρέπει ε, να έχει το δικαίωμα καταναλωτής να προστατεύεται, να μην είναι παραπλανητική διαφήμιση ενός προϊόντος. Και αυτά λοιπόν τα προφίλ της διατροφικής αξίας ενός τροφίμου είναι παραπλανητικά, γιατί δεν στέκουν. Και επιπλέον, επιπλέον λέγω, είναι και άχρηστα αυτά. Ε, για να αξιολογήσει κανείς κατά πόσο είναι σωστοί οι ισχυρισμοί, αν αληθεύουν ή όχι αυτοί οι ισχυρισμοί για την υγεία. Ανεξάρτητα από το γεγονός αν ε, έχει ε, ο ζάχαρη, λίπος ή αλάτι ένα τρόφιμο. Να αποφασίζει ο καταναλωτή τι θέλει. Δεν θα του πούμε ποιο τρόφιμο είναι καλό ή κακό. Βεβαίως θα πρέπει να είναι η κακο Βεβαίω διαφάνεια. Γι' αυτό η τα κατάταξη αυτή η προκατακτική είναι άχρηστη. Δεν μπορούμε εμεί να λέμε αυτό είναι καλό τρόφιμο και το άλλο είναι κακό. Και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Έχω και μια ερώτηση για την ΕΦΣΑ και τις διαφημίσεις που γίνονται. Έχει ε, καθυστερήσει πάρα πολύ, 1,5 χρόνο περίπου περιμένουμε να γνωμοδοτήσει η ΕΦΣΑ και θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα χρόνο, για να μην πω και παραπάνω, ε, ίσως και 1,5, για να δώσει τον κατάλογο των επιτρεπωμένων ε, δηλώσεων στη διαφήμιση για θέματα υγείας. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο και ε, διακόπτη. Μια σταδιακή ε, δημοσίευση των στοιχείων. Ε, αυτό όμω είναι παραπλανητικά. Κύριε Σπανιό. Κύριε Επίτροπε, τρία σημεία θέλω να θίξω. Πρώτον, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της γρήπης. Κάθε φορά που ασχολείστε με το θέμα μιλάτε για πανδημία. Όλοι γνωρίζουν τώρα σε όλο τον κόσμο ότι ήταν μια επιδημία η οποία ήταν πολύ λιγότερο θανατηφόρος από μια απλή εποχιακή γρήπη. Οπότε είναι σωστό νομίζω όταν μια επίσημη αρχή όπως εσείς αναφέρετε στο θέμα αυτό να χρησιμοποιεί τους σωστούς όρους, τους όρους που είναι αντίστοιχοι με τα διαπιστωθέντα. Όπως ακριβώς διευκρινίσατε, πάρα πολύ σωστά άλλωστε, το θέμα της διαχείρισης αυτής της κρίσης, έτσι όπως τη βιώσαμε, κινδυνεύει ε, στο να δημιουργήσει αμφιβολίες στον πληθυσμό για τις μελλοντικές πανδημίες. Γιατί από ό,τι φαίνεται δυστυχώς κάποια στιγμή θα υπάρξουν τέτοιου είδους πανδημίες στο μέλλον. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να προσπαθήσουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως το είπε η κυρία Ρεβαζή και όπως το είχε πει και ο κύριος Μπαρόσο παλαιότερα να υπάρχει η δυνατότητα ένα όργανο διεθνές να μπορεί να διασφαλίζει ουσιαστικά τους Ευρωπαίους για τους κινδύνους τους οποίους διατρέχουν και για το τι πράγματι συνέβη. Άλλο θέμα, η ενημέρωση των ασθενών. Υπήρξε μια ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε εμπλεκομένους και εσάς και τον κύριο Λάινεν φυσικά και δεν κατανοώ κύριε Επίτροπε τη θέση σας από τη μία θέλετε να πάμε πιο μακριά, ακόμα παραπέρα στην ενημέρωση των ασθενών και στην, στον ανεξάρτητο ρόλο των ομάδων των Χριστών, των συλλόγων των Χριστών, ενώ από την άλλη η οδηγία την οποία προτείνεται δεν θα το επιτρέψει αυτό. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα εδώ και χρήζει διευκρίνηση στη συγκεκριμένη θέση σας. Ευχαριστώ. Ρίχαρτ απουσιάζει αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Τρεμόπουλος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα επανέλθω ε, κύριε Επίτροπε στο θέμα των ε, γενετικά τροποποιημένων. Υπάρχει ένα αίτημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Βιοκαλλιεργητών για ένα νέο ευρωπαϊκό μορατόριο όσο αφορά την έγκριση και καλλιέργειά τους μέχρι να εκπληρωθούν οι απαιτήσει που είχαν θέσει οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Περιβάλλοντος το Δεκέμβριο του 2008. Μιλήσατε για την επιστήμη και ότι σέβεστε. Ε, την ίδια στιγμή έχουμε μεροληπτική στάση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων, την ΕΦΣΑ, η οποία παρόλο το ανεξάρτητη αρχή φαίνεται να ταυτίζεται με τις θέσεις των εταιριών βιοτεχνολογίας. Επίσης, η δυνατότητα των κυβερνήσεων να απορρίπτουν τις ε, τροποποιημένες γενετικά καλλιέργειες στις χώρες τους δεν αρκεί για να δικαιώσει τη νέα πολιτική της Κομισιόν να δίνει απλόχερα εγκρίσεις για όποια νέα ποικιλία ζητούν οι εταιρείες ανεξάρτητες επιστημονικές έρευνες αμφισβητούν την αμεροληψία της εφσα ε, και τονίζουν τα σοβαρά προβλήματα διαφάνειας που εμποδίζουν τη διασταύρωση των πορισμάτων από την επιστημονική κοινότητα. Εταιρείες βιοτεχνολογίας έχουν ε, λάβει γνώση εμπιστευτικών πορισμάτων πριν από την κοινωνία των πολιτών και ανώτερα στελέχη της έχουν μεταπηδήσει σε υψηλόβαθμες θέσεις εταιριών βιοτεχνολογίας η ίδια η εφσα δηλώνει αδυναμία να μελετήσει τις μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων. παρ' όλα αυτά εσείς η επιτροπή στηρίζεστε αποκλειστικά στις γνωμοδοτήσεις της. ρωτώ με λοιπόν ε, υπάρχει συγκεκριμένη ε, προσπάθεια να αξιολογηθεί η κριτική αυτή για την αξιοπιστία της ε, της ΕΦΣΑ και με τι διαδικασίες προλαμβάνετε ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων τέλος γνωρίζετε αυτή τη διακήρυξη και το αίτημα για μορατόριουμ στην καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων. Σκοπεύετε να το αποδεχθείτε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η Καρίν Κάδο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η ναι, κυρία Κάλμπαχ, ακούσαμε ε, πόσο ευρία είναι η παλέτα των θεμάτων που χειρίζεστε. Και μιλήσαμε για την πανδημία της ε, γρήπης ΙΤΑ 1 ή 1. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την ανασωποίηση, πιο συγκεκριμένα. Διαπιστώσαμε ότι στην Ευρώπη, κυρίως στα παιδιά ε, και σε ενηλίκους όμως, μειώνεται ο εμβολιασμό. Και μεταξύ αυτών, γιατί ορισμένες ε, ασθένειες όπως είναι η λαρά, οι μαγουλάδες, η παροτίτιδα, ε, τα εμβόλια που κάναμε εμείς όταν ήμασταν μικροί έχουν μειωθεί οι ασθένειες και ο κόσμος δεν θέλει να εμβολιάζει τα παιδιά του. Έχουμε όμως και τουρισμό ε, ανοιχτά σύνορα και ε, ξαναεμφανίζονται αυτά τα νοσήματα που θεωρήσαμε ότι είχαν απομακρυνθεί από την Ένωση. Τι θα γίνει λοιπόν με ε, τα προγράμματα τα εμβολιαστικά των κρατών μελών που είναι διαφορετικά μεταξύ τους για να ανοσοποιούνται τα παιδιά μας στην Ευρώπη όλο και περισσότερο ξανά όπως και στο παρελθόν. Αν θέλετε να απαντήσετε παρακαλώ. Cross-border healthcare Um, η διασυνοριακή υγεία είναι κάτι για το οποίο έχουμε συνομιλήσει με την Ισπανική Προεδρία. Και συζητήσαμε και την πρόταση που αναφέρατε της Προεδρίας. Στην τελευταία συνεδρίαση των Υπουργών Υγείας ακούστηκε η πρόταση για μια μελέτη που νομίζω ότι περιέχει τα στοιχεία πιθανής συμφωνίας μέχρι τον Ιούνιο. Οπότε και θα σας έρθει η πρόταση για δεύτερη ανάγνωση. Ίσως είμαι υπεραισιόδοξος, αλλά νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή τέτοια πιθανότητα. Για τη δημόσια υγεία συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη έρευνα για τις επιπτώσεις του ινοπνεύματος και άλλων τέτοιων ουσιών που βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία είναι τομέα στον οποίο επίσης πρέπει, με τον οποίο πρέπει επίσης να ασχοληθούμε αλλά πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχουν πολλοί περιορισμοί και φραγμοί στη δραστηριότητά μας θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε ώστε να μην περιοριστούμε στην έρευνα αλλά και σε καμπάνιες πληροφόρησης και αποτροπής. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερες καμπάνιες αποτροπής. Αυτό μπορεί να το κάνει η Κομισιόν. Και έτσι η υγεία να καταντήσει βιώσιμη για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις ζημίες. Για τις ε, αναλύσεις των συστατικών σας είπα, εμείς βασιστήκαμε σε επιστημονικά δεδομένα της ΕΦΣΑ και κάναμε μια μισούλα αλλά πρέπει να αποσαφηνίσω το εξής. Οι αναλύσεις αυτές δεν θα ισχύουν παρά μόνο από τη στιγμή που έχει γίνει αποδεκτή μία μάρκα ή κάποιο τρόφιμο καινούριο και θα αρχίσουν να ισχύουν διατάξεις μόνο αν παραβιάζει τα ανενομισμένα ποσοστά. Αυτό είναι δίκαιο και λογικό και για τους καταναλωτές και καταναλώτριες. Για τη γρήπη ή τα έναν ή ένα τι να σας κάνω, πανδημία την είπανε. Τους πρώτους δε μήνες της υπήρξε γρήγορη αντίδραση και εμβολιασμό με ρυθμούς πολύ πιο γρήγορους από οτιδήποτε είχε ποτέ ξαναγίνει αναλόγως. Μάλιστα μία από τις ε, ένας από τους λόγους της χαμηλής θνησιμότητας της γρήπης αυτής μπορεί να οφείλεται στους εμβολιασμούς. αν δεν είχαμε εμβολιάσει και αν είχαμε θεωρήσει τη γρήπη αυτή ως κανονική μπορεί να ήταν πολύ χειρότερα τα αποτελέσματα. Αυτό πρέπει να αναλύσουμε λοιπόν για να είμαστε βέβαιοι ότι ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα με τον αντικειμενικότερο τρόπο. Δυστυχώς συμφωνώ, ο εμβολιασμό θεωρήθηκε άχρηστος από όλο και περισσότερους ανθρώπους, ενώ τώρα βλέπουμε ότι στη Βουλγαρία, παραδείγματο χάρη την περασμένη εβδομάδα, ξέσπασε γρήπη. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να επιμένουμε για τον εμβολιασμό και ότι είναι τρόπος αντιμετώπισης των ασθενειών για την πληροφόρηση των ασθενών. Τι να σας πω, ακούμε αυτά που μας λέτε και θα θέλαμε το Κοινοβούλιο να συνεχίσει τις συζητήσεις του. Ήδη σημειώσαμε ορισμένα στοιχεία τους και τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί που κατ' εμέ είναι πολύ λογικές και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή και με τις υπόλοιπες τροπολογίες της δικές σας για το θέμα αυτό. Τέλεια. Η Κατερίνα Σουλή. Ευχαριστώ Και Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, τεράστιες οι ευθύνες σας. Σημείωσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι σας απασχολεί η ευημερία των ζώων που καλύπτεται από το άρθρο 13 που λέει ότι η κοινότητα και τα κράτη-μέλη λαμβάνουν υπόψη τους τα κριτήρια για την ευημερία των ζώων. Τι προβλέπετε να κάνετε λοιπόν ως Επίτροπος υπεύθυνο για την υγεία για να διασφαλιστούν οι στόχοι αυτή της ευημερίας των ζώων και πιο συγκεκριμένα για την έρευνα και τις δοκιμές για τα καλλιντικά Αντίθετα από την ιατρική έρευνα, η έρευνα αυτή μπορεί να γίνει και χωρίς ζωικές δοκιμές. Και υπάρχει η οδηγία για τα καλλιντικά που μιλάει για τις δοκιμές αυτές. Τι πρόκειται να γίνει. Ευχαριστώ πολύ ο Μάριος Πουρή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο Ντάλι. Θα ήθελα να μάθω αν έχετε στο πρόγραμμά σας πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία. Είναι μια μεγάλη μάχη η οποία δίνεται κάθε χρόνο, μεγαλώνει η μάχη αυτή και γι' αυτό θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Μήπως θεωρείτε ότι στα θέματα της ψυχιατρικής δεν θα πρέπει να δοθούν περισσότεροι πόροι στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογίας. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα διαφέρουν από χώρα σε χώρα και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αρκετή πρόοδος αλλά υπάρχουν και πολύ σημαντικές ασυγχώρητες καθυστερήσεις. Αγιούσο. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε για τις εξηγήσεις και το πρόγραμμά σας. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε καλό επίπεδο, πολύ καλό επίπεδο προστασίας της ασφάλειας των τροφίμων και έχουμε και πολύ αυστηρή νομοθεσία και τα κράτη μας ενισχύουν ε, την νομοθεσία της Ευρώπης. Αλλά όλα αυτά που τρώμε δεν παράγονται όλα στην Ευρώπη. Εισάγουμε τρόφιμα που δεν τηρούν τους ίδιους κανόνες. Γιατί ο ΠΟΕ δεν μας επιτρέπει να ε, απαγορεύσουμε την είσοδο αυτών των προϊόντων και εμείς δεν τα ελέγχουμε. Ούτε στην παραγωγή, ούτε στην κατανάλωση, ούτε στην προέλευση. Και αν έχετε χρόνο να μιλήσουμε για τις κονσέρβες ψαριών που εισάγουμε από την Νοτιοανατολική Ασία. Έχετε καμιά πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και για τα κλωνοποιημένα ζώα. Ψηφίσαμε να αποσυρθεί από την πρόταση Novel Food ε, αυτή η ρυθμισή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας καταθέσει νέα πρόταση που να απαγορεύει τη χρήση χρονοποιημένων ζώων για την παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης. Μπορεί να το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας καταθέσει πρόταση να απαγορεύει δηλαδή την παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης από κλωνοποιημένα ζώα. Και μπορούμε να ξέρουμε ποια ζώα είναι κλωνοποιημένα. Αυτό διαπιστώνεται. Αν δεχτούμε λοιπόν ότι πρέπει αυτό να απαγορευτεί, μετά πώς θα το ελέγξουμε στα τρόφιμα. Μπορούμε να το απαγορεύσουμε στην Ένωση, αλλά θα μας έρθει έξωθεν. Τι λύση έχετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Και τελευταίο. Έχω και τελευταίο. Δεν τέλειωσα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Αναφερθήκατε επανειλημμένα στις διασύνοριακές υπηρεσίες υγείας και στην οδηγία την αντίστοιχη. Ήμουν ονομοδότρια στην έκθεση για την εσωτερική αγορά και στην έκθεση πρωτοβουλίας μου αρχικά είχα ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη την πραγματική πρόκληση που θα αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια, τη γύρανση δηλαδή του πληθυσμού και τα, την ειδική φροντίδα που θα πρέπει να δοθεί στον πληθυσμό, τον ευρωπαϊκό, ο οποίος κινείται και μετακινείται εκτός συνόρων. Η Ισπανική Προεδρία είναι σαφής γύρω από το θέμα αυτό, δεκτική. Ο προκάτοχός σας στηρούσε στάση αναμονής. Εγώ νομίζω ότι το θέμα αυτό παρόλα αυτά είναι κατεπήγον. Θα εμπλουτίσετε το κείμενό σας μέσω αυτής της προβληματικής, γιατί έχουμε να κάνουμε με υπηρεσίες υγείας που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, βοηθούν την περιφερειακή συνοχή και συνοδεύουν κοινωνικά πληθυσμούς οι οποίοι αυξάνονται συνεχώς. Ευχαριστώ, Κρήτον. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε. Επίτροπε, οι πολίτες ανησυχούν από την πρώτη αυτή έγκριση ε, ΜΚΟ στην Ευρώπη. Από το 1998 είναι η πρώτη που ε, επιτρέπεται. Λέτε ότι οι αποφάσεις ε, βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Και βεβαίως τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι αξιόπιστα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι πήρα την απόφαση για την πατάτα φλόρα ε, μετά από θετικές επιστημονικές υποδείξεις. Έχει δύο όμως μελέτες από την ΕΦΣΑ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι γεγονός αυτό, αλλά είναι επίσης γεγονός ε, ευρέως ε, διαδεδομένο ότι οι μελέτες αυτές θεωρούνται μη αξιόπιστες. Και τότε ζητήθηκε και τρίτη μελέτη, όχι μόνο από την ΕΦΣΑ, αλλά και από κάποιον άλλον. από την ΕΜΕΑ. Λοιπόν, ε, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ζήτησε νέα μελέτη εφόσον αυτές θεωρούνται αναξιόπιστες. Ευχαριστώ, η Άνια Βάισκερβερ. Ευχαριστώ. Έχω τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ε, πρώτον, για τις ε, Απομιμή ε, πραγματική απάτη και ε, παραπλάνηση του καταναλωτού. Ε, σας ερωτώ, τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια είναι η κατάσταση των Σα ερωτω τι γινεται στην ευρωπαικη επιτροπη ποια ειναι Η Επιτροπή Περιβάλλοντος σαφέστατα ήταν υπέρ. Ακούω λέτε, λένε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα νομικό με τη λέξη imitate, τι θα πει, ότι απομίμηση. μπορούμε να το βρούμε αλλιώς. Ε, να το πούμε αλλιώ. δηλαδή υπάρχουν προϊόντα που είναι ε, ανάμειξη φυτικών ε, λοιπόν και το πουλάνε για τυρί. Μετά, για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, το συζητήσαμε και προηγουμένω Χαίρομαι που ο πρόεδρος Μπαρόσο το δηλώνει και εσείς υποστηρίξετε να αποφασίζουν τα κράτη-μέλη εάν θα καλλιεργήσουν μεταλλαγμένα ή όχι. Αυτά τα σχέδια τα έχετε συγκεκριμενοποιήσει και σε ποιο βαθμό. Και τι γίνεται με τι περιφέρειες. Μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν οι περιφέρειες στο εσωτερικό των κρατών μελών. Αυτό βέβαια νομικά ε, πρέπει να ρυθμιστεί από τα κράτη-μέλη, αλλά θέλω να μάθω αν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό. Και για τον ασθενή, και εγώ είμαι υπέρ του χειραφετημένου ασθενού και, του ενημερωμένου ασθενού. Να γνωρίζει ε, μια πλατφόρμα, α πούμε, ε, στο διαδίκτυο να δημιουργηθεί που να είναι και ε, ουδέτερη και να ελέγχεται ανεξάρτητα για να ενημερώνεται ο ε, για μεθόδους θεραπείας, για φάρμακα, για ασθένειες. Ε, και αυτό έχει ήδη εγκριθεί στην Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτού και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα το εγκρίνουμε. Έχω επαφές με την Κομισιόν. Εσείς τι λέτε προσωπικά γι' αυτό. Ευχαριστώ. Παρβάνοβα. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο. Τρεις σύντομες ερωτήσεις. Τρεις ερωτήσεις, χιλιάδες ίσως οι απαντήσεις. Καταρχάς, ο γυράσκον πληθυσμός και η κρίση που δημιουργείται εξ αυτού στα συστήματα υγείας. Θέλετε να ζητήσετε από τα κράτη-μέλη να προετοιμάσουν καλύτερα την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει φυσικά άμεσες συνέπειες στη διαχείριση των συστημάτων υγείας. Καταρχάς, η λεγόμενη ηλεκτρονική υγεία, το e-health, τι σκοπεύετε να κάνετε προς την κατεύθυνση αυτή. Έχετε επίσης ε, περαιτέρω ιδέες ή προτάσεις για τις κλινικές δοκιμές των φαρμακευτικών ουσιών. Ευχαριστώ. Μπελιέ, τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ντάλη. Μιλήσαμε αρκετά για τα γενετικά τροποποιημένα σήμερα και είναι ευθύνη όλων μας να διασφαλίσουμε στο σύνολο των Ευρωπαίων μια αποτελεσματική και εναρμονισμένη ανταπόκριση στις ανησυχίες τους ιδιαίτερα με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Μία ευχή λοιπόν να εκφράσω και μετά μια ερώτηση. Καταρχάς, θα ήθελα να επιστήσω ακόμα μια φορά την προσοχή σας για τα θέματα της διαφάνειας και πρόσβασης στην πληροφορία και σχετικά με τις επιστημονικές αξιολογήσεις τις οποίες κάνει το ΕΦΣΑ και για την ετικετοθεσία των προϊόντων που μπορεί να περιλαμβάνουν ε, γενετικά τροποποιημένα. Γι' αυτό ακριβώς σήμερα το πρωί ε, κάναμε μια πρόταση μέσω της ψηφοφορίας μας σχετικά με το κρέας το οποίο καταναλώνουν ε, είναι το ελάχιστο το οποίο ζητάμε και γι' αυτό η Επιτροπή σας θα πρέπει να ενταποκριθεί στα προβλήματα που υπάρχουν σε επίπεδο ετικετοθεσίας. Για τις επιστημονικές αξιολογήσεις είπατε ότι βασίζεται τις αποφάσεις σας ακριβώς σε συγκεκριμένες επιστημονικές μελέτες. Αναγνωρίζεται όμως από την ίδια την ΕΦΣΑ ότι οι επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει για τα γενετικά τροποποιημένα δεν περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των κινδύνων. Αγνοούν κάποιες αντιθετικές, αν θέλετε, μελέτες επιστημονικές που έχουν κάνει εξωτερικοί οργανισμοί. και δεν έχουμε την δυνατότητα εμείς να έχουμε τα συστήματα και τα πρωτόκολλα ελέγχου που θα μας επιτρέψουν να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των αξιολογήσεων. Λόγω ακριβώς αυτής της έλλειψης κοινωνικονομικής ε, μορφής ελέγχου δημιουργούνται προβλήματα για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Διαρωτώ με λοιπόν κύριε Ντάλη Ποιες είναι οι συνθήκες για την Επιτροπή σας της εφαρμογής της αρχής της πρόληψης. Καταλάβαμε την ερώτησή σας, λέει ο κ. Κάντε το ίδιο που έκανε ο Ποτότσνη. Μπορείτε γραπτά να δώσετε απαντήσεις αν δεν προλάβετε να απαντήσετε σε όλες. Τρία-τέσσερα λεπτά μόνο έχετε στη διαθεσή σας και στις υπόλοιπες γραπτά. για τα φαρμακευτικά προϊόντα και την αξιολόγησή τους. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητά τους και όχι μόνο την ασφάλειά τους. Η γύρανση του πληθυσμού είναι βασική μου προτεραιότητα την επόμενη πενταετία. Είναι η βάση επί της οποίας θα πρέπει να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας Η γύρανση με υγεία είναι θα έλεγα βασικό στόχος αυτής της περίοδου. Και όχι μόνο με υγεία αλλά και παραγωγική γύρανση. Γιατί πρέπει κανείς να είναι υγιής για συγκεκριμένους λόγους και όχι απλά να μην κάνει τίποτα. Και εδώ έρχεται και η ηλεκτρονική υγεία. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο θέμα της γύρανσης. Χαίρομαι που η Ισπανική Προεδρία στα πλαίσια της αναθεώρησης της διαμεθοριακής πρωτοβουλίας κάνει συγκεκριμένε προτάσεις. Θέλουμε όλους να έχουμε μια πιο συντονισμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων της ηλεκτρονικής υγείας, e-health. Είναι κάτι, εν πάση περιπτώσει, το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουν τα συστήματα να λειτουργήσουν σωστά για την ενημέρωση των ασθενών. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την πρόταση που προήλθα από την Επιτροπή ΕΝΒΗ για τη δημιουργία ενός πόρταλ το οποίο θα λειτουργήσει σαν φίλτρο ανάμεσα στις ε, φαρμακευτικές εταιρείες που οφείλουν να δώσουν τις πληροφορίες και τους ασθενείς οι οποίοι θα πρέπει να προστατεύονται από το μάρκετινγκ των φαρμακευτικών ουσιών. Και αυτό θα βοηθήσει να κρατήσουμε ικανοποιητικά ε, επίπεδα προστασίας για τα γενετικά τροποποιημένα και για τα υπόλοιπα θα απαντήσω ε, γραπτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους γενικές δηλώσεις ότι η έλεγχη αυτή δεν είναι αξιόπιστη κτλ. Το ΕΦΣΑ ελέγχεται από τα όργανα και αν υπάρχουν θέματα με το ΕΦΣΑ θα πρέπει να τους τα αναφέρουμε για να τα αναλύσουν. Εγώ έχω επισκεφθεί την ΕΦΣΑ πρόσφατα και είδα ότι θα έπρεπε να έχουμε μια πιο μόνιμη ελεγκτική λειτουργία σχετικά με την ανεξαρτησία των γνωμοδοτήσεων οι οποίες περνούν από τις διάφορες επιτροπές που λειτουργούν στο εσωτερικό του συστήματος του ΕΦΣΑ. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να ενισχύσουμε την οργάνωση αυτή και όχι να την δαιμονοποιούμε όταν οι αποφάσεις της δεν μας αρέσουν. Ευχαριστώ Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση των ιδεών σας και για την απάντηση στα περισσότερα από τα ερωτηματικά που τέθηκαν.